Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί βραβευθέντες Ζαχάροφ. Ε, άρχεται η συνεδρίασή μας. Σήμερα είναι ε, μια σημαντική στιγμή. Το 2011 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά της Αραβικής Άνοιξης. Ε, είναι τιμή για μένα να... Ε, απονείμω το βραβείο Ζαχάροφ στην Ελευθερία Σκέψης του 2011 σε πέντε θαραλέες γυναίκες και θαραλέους άντρες που αντιπροσωπεύουν αυτή την Αραβική Άνοιξη. Το βραβείο απονέμεται στους κυρία Ασμά Μαχβούζ από την Αίγυπτο. τον κύριο Αχμέτ Αλσανούση από τη Λιβύη. την κυρία Ραζάν Ζάι από τη Συρία. Τον κύριο Αλή Φαρζάτ από τη Συρία. Και τον εκλειπώντα Μοχάμετ Μπουαζίζη από την Τινησία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια. Όλοι ε, θεωρούμε ότι η ελευθερία σκέψης, η ανθρώπινη εξυπρέπεια και η ελευθερία έκφρασης ε, είναι σημαντικά αγαθά, όπως επίσης ε, και η ε, χρηστή διακυβέρνηση με την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στους ε, πέντε ακτιβιστές της Αραβικής Άνοιξης. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τις προσπάθειες όλων όσοι αγωνίζονται για αξιοπρέπεια, θεμελιώδεις ελευθερίες ε, και πολιτική αλλαγή στον αραβικό κόσμο. Ανατρέχοντας στα γεγονότα του, έτους, του τρέχοντος έτους, μετά την Επανάσταση στην Τινησία, γίναμε μάρτυρες της ε, ε, πτώσης της δικτατορίας και των ελεύθερων αλλαγω, ε, εκλογών. Γι' αυτό το λόγο απονείμαμε και το βραβείο Ζαχάροφ στον εκλειπώντα Μοχάμετ Μποαζίζη, έναν νέο μικροπολιτή, έναν νεαρό μικροπολιτή, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε αφού οι αρχές της ε, χώρας του επανειλημμένως του αρνήθηκαν τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα αξιοπρέπειας. Από τότε η, ιστορία σάρωσε τη Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή. Σε πολλά μέρη αυτός ο αγώνας ακόμα συνεχίζεται τώρα που μιλάμε. Στη Συρία για παράδειγμα ε, η, ε, όσοι διαμαρτύρονται αντιμετωπίζονται με δακρυγόνα, ε, σφαίρες, τάγκς, ε, κρατήσεις, συλλήψεις και βασανιστήρια. Οι, ε, νεκροί ξεπερνούν τους 5.000, μεταξύ αυτών και 300 περίπου παιδιά. Για να τιμήσουμε και να θυμηθούμε τον κύριο Μπουαζίζη και όλους αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον αγώνα στον αραβικό κόσμο, θα ήθελα να ζητήσω από όλους εμάς ένα λεπτό σιγής. Τα ιστορικά γεγονότα μας υπενθυμίζουν επίσης και τις ευθύνες μας συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης υποστήριξης ε, της ε, ε, κοινωνίας των πολιτών. Μεταξύ ημών έχουμε δύο νέες γυναίκες που αντιπροσωπεύουν αυτή ακριβώς τη νέα γενιά την Ασμα Μαχβούς και την Ραζάμ Ζάιτουνεχ από την Αίγυπτο και τη Συρία αντίστοιχα. που αγωνίζονται όχι μόνο για σεβασμό αλλά και για καλύτερες ε, προοπτικές για το μέλλον. Οι, οι γυναίκες έπαιξαν ένα αποφασιστικό ρόλο στην Αραβική Άνοιξη και ελπίζω ότι η θαραλέα τους συνεισφορά, η θαραλέα τους συμμετοχή αποτελεί ένδειξη ότι οι πολιτικές αλλαγές θα φέρουν βελτίωση και στην κατάσταση και τα δικαιώματα των γυναικών σε αυτή την περιοχή. Σήμερα καλωσορίζουμε μια νέα και σημαντική γυναίκα, την Ασμά που κινητοποίησε τους Αιγύπτιους να βγουν στο δρόμο, στη Μιλατεία Ταχρήρ και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα και σύμβολο του πώς ε, ένας άνθρωπος ε, μπορεί να κάνει τη διαφορά με την έμπνευσή του και με την πεποίθησή του παρόλα τους ε, κινδύνους και την, τον εκφοβισμό εκ μέρους των αρχών. Κυρία Μαχβούς, θα ήθελα να σας καλέσω να λάβετε το λόγο. The podium beneath, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και σας ευχαριστώ όλους για την υποδοχή σας και για την απονομή αυτής ε, της ανταμοιβή που είναι μια ανταμοιβή της Αραβικής Επανάστασης και αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής για την Ευρώπη και για τον αραβικό κόσμο και για την αμοιβαία κατανόηση επί μεγάλο χρονικό διάστημα ζήσαμε πάνω σε στερεότυπα που χωρίζουν τον κόσμο. Τώρα που έχει στραφεί το ενδιαφέρον στον αραβικό κόσμο, όλοι είδατε ότι μπορείτε να είστε υπερήφανοι για τον αραβικό κόσμο. Ο αραβικός κόσμος έχει κατά νου τις ε, αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρήνης. Και ε, αυτή η τιμή που γίνεται είναι τιμή προς τους ήρωες της Επανάστασης. Είναι μια τιμή προς όλους τους νέους Αιγυπτίους, νέοι που θυσίασαν τη ζωή τους, που είναι πιο θαραλέοι από μένα. Θυσίασαν τη ζωή τους, θυσίασαν τα πάντα για την ελευθερία, για την επανάσταση. Η Αιγυπτιακή Επανάσταση επέτρεψε την πτώση του καθεστώτος παρά την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών ευρωπαϊκών κρατών, υποστήριξη που διδόταν στον ε, Μουμπάρακ πριν την Επανάσταση. Υπάρχουν ε, πολλά για τα οποία χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να μπορέσει να αλλάξει το καθεστώς. Τα καθεστώτα δεν βασίζονται σε ένα άτομο, βασίζονται στην υποστήριξη πολλών ατόμων. Και είμαι υπερήφανη που υποστηρίζω τον ε, Αιγυπτιακό λαό που κατέληξε σε τόσες επιτυχίες βασιζόμενοι στην βασιζόμενος ε, στην ειρηνική ε, πάλι. Το καθεστώς Μουμπάρακ δεν έχει πλέον υποστήριξη και οι παλαιοί υποστηρικτές όπως ε, το Στρατιωτικό Συμβούλιο δεν θα επιτύχει. Υπάρχουν νέοι που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για τους στόχους της επανάστασης και για την αναγέννηση ενός μη στρατιωτικού κράτους που θα προστατεύει τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες. Κάθε φορά που απειλείται μια ανθρώπινη ζωή, θα πρέπει να υπάρχει μια ταχεία αντίδραση. Γιατί να πρέπει να περιμένουμε μετά τη δολοφονία ανθρώπων, μετά τη δολοφονία πολλών ανθρώπων για να αναλάβουμε δράση. Αρκεί μία δολοφονία, αρκεί μία παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ελπίζω ότι η πρώτη προτεραιότητα σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι να δώσουμε στους ανθρώπους τα δικαιώματά τους για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον κόσμο στον οποίο όλοι προσβλέπουμε. Εν κατακλείδη θα ήθελα να σας μεταφέρω το θαυμασμό μου για όλους τους μάρτυρες της Αραβικής Επανάστασης. Δεν θα προδώσουμε όλους αυτούς. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το όνειρο, το όραμα της αλλαγής. Δόξα λοιπόν στους μάρτυρές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Η άλλη νεαρή βραβευμένη, την οποία ανέφερα, είναι η Ραζάν Ζάι Τούνεχ. Ε, είναι αναγκασμένη να κρύβεται. Δεν είναι μαζί μας σήμερα. Όμως συνεχίζει να καταγγέλει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του blog της παραβιάσει εκ μέρου των Συριακών αρχών. Αυτό δείχνει το εξαιρετικό της κουράγιο και θάρρος. Μας ε, έστειλε ένα συγκινητικό γραπτό μήνυμα. Ένα μήνυμα ελπίδας για μια ε, ελεύθερη και πολυφωνική Συρία. Το μήνυμα αυτό σας έχει σταλεί, συνάδελφοι. Σα εστάλει σήμερα το πρωί. Έχουμε όμως μαζί μας έναν άλλο τιμηθέντα με το βραβείο Ζαχάροφ που είναι ο Αχμέτ Αλσανούση. Είναι ένα από αυτά τα εξαιρετικά άτομα που προσπάθησαν να ρίξουν ε, ένα δικτάτορα εδώ και πολύ καιρό και πλήρωσε βαρύ το τίμημα της προσπάθειάς του. Ε, είναι ο άνθρωπος που έμεινε πιο πολλά χρόνια ε, κρατή ε, για ε, ε, στην, για 31 συγκεκριμένα χρόνια κρατήθηκε στη Λιβύη. Είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνο για τους πολιτικούς κρατούμενους του Εθνικού Συμβουλίου της Λιβύης. τα δεινά που έζησε ελπίζω ότι θα βραβευθούν με την εθνική ε, συμφιλίωση στη Λιβύη. Η εμπειρία του νομίζω ότι θα χρησιμεύσει πολύ σε αυτή τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης. Κύριε Αλσανούση, θα ήθελα να πάρετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας χαιρετίζω θερμά και συνάμα σας ευχαριστώ και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την επιλογή σας ε, και για ε, ότι μου απονείματε το βραβείο Ζαχάροφ. Αυτό είναι μια, αυτό είναι μια χειρονομία που πραγματικά ενθαρρύνει τον ε, λαό της Λιβύης, λαός της Λιβύης ο, οποίος με συνεχάρει για την απονομία αυτού του βραβείου αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την ε, προάσπιση των ε, ελευθεριών στην ε, Λιβύη, τη δημοκρατία και ένα καθεστώς το οποίο θα βασίζεται στην ισοτιμία όλων των πολιτών της όπου οι γυναίκες θα μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την ψήφο τους και θα εισακούεται η φωνή τους διότι οι γυναίκες ε, πραγματικά θυσιάστηκαν. Η γυναίκα θυσίασε την ζωή της, τα παιδιά της, τους συγγενείς της προκειμένου να πετύχουμε τους ε, στόχους, δηλαδή να απαλλαγούμε από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ε, το οποίο μας οδήγησε σε αποκλεισμό για 42 χρόνια στην ταπείνωση στην... όλα αυτά τα χρόνια μας ε, οδήγησαν σε μια απομόνωση από τις υπόλοιπες κοινωνίες Οι γυναίκες με μόνο όπλο τις πεπιθήσεις τους και τη βούλησή τους μπόρεσαν ε, να κάμψουν το καθεστώς αλλά φυσικά με την στήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το, το οποίο θέλαμε να εκφράσουμε την ε, ευγνωμοσύνη μας. Προσβλέπουμε στην ανοικοδόμηση της ε, χώρας μας και στη δημιουργία μιας κοινωνίας ανεκτικής ακόμα και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι διάπραξαν εγκλήματα κατά των αδελφών μας ε, Άνθρωποι οι οποίοι κατέθεσαν τα σπίτια μας παρακολουθούσατε μέσω από τις τηλεοράσεις και από τις δορυφορικές εκπομπές όλες τις παραβιάσεις που γνώρισε η Λιβύη. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη, την οικονομική, τη διπλωματική αλλά και τη στρατιωτική που μας παρήχατε. Ήμασταν ένας λαός άοπλος και ο δικτάτορας ήθελε να μας υποτάξει με την βία και την ισχύ μέσω των σχέσεων που είχε δημιουργήσει και αναπτύξει τα τελευταίο καιρό ε, κάποια άλλα κράτη κράτη που τον στήριζαν για ποικίλου λόγους, για λόγους οικονομικούς και άλλους. Αλλά όλα αυτά τα έθνη, όλα αυτά τα κράτη ε, αντελήφθησαν ότι η νίκη θα είναι με την πλευρά του Λιβικού λαού. Ευχαριστούμε λοιπόν την Ευρώπη για τις θέσεις της και για τις πράξεις της. Ευχαριστούμε και την διεθνή κοινότητα, αλλά θα πρέπει να ομολογήσουμε πως οι Ευρωπαίοι ήταν οι πρώτοι που στήριξαν τον άοπλο Λαό μας. Και χάρη σε αυτήν την υποστήριξη των Ευρωπαίων μπορέσαμε να απαλλαγούμε από ένα δικτατορικό καθεστώς που δίκησε 42 χρόνια. Ε, φυλάκισή μου και να θέσει τέλος και στην ε, φυλάκισή μου η οποία δίκησε 31 χρόνια συμπεριλαμβανομένων 9 ετών σε απομόνωση, σε κελί απομόνωσης όπου και βασανίστηκα δεν ε, τύχανα ιατρικής περίθαλψης αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν έχασα την ελπίδα μου θέλουμε να συνεχίζουμε να ζούμε με την διεθνή κοινότητα και να την χάνουμε ισότιμης αντιμετώπισης. Δεν θέλουμε να μας περιγράφουν πλέον σαν κράτος του τρομοκρατών. Εμείς αγαπάμε τη ζωή και επίσης σεβόμεθα τη ζωή των συναδέλφων μας. Ελπίζουμε αυτό το βραβείο Ζαχάροφ να μας επιτρέψει να πετύχουμε περαιτέρω πρόοδο, όχι μόνο εμείς, αλλά και τα υπόλοιπα κράτη τα οποία ε, γνωρίζουν δικτατορίες. Ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει για να ε, επιτύχουμε τους στόχους μας. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, αλλά χάρη στην υπομονή μας και την αίμονή μας μπορέσαμε να πετύχουμε και φτάσαμε στο να έχουμε ένα νέο σύνταγμα το οποίο ψήφισε ο λαός. Ειρήνη Ημίνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το βραβείο Ζαχάροφ απονέμεται για την ελευθερία σκέψης και η ελευθερία σκέψης μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Μερικές φορές ε, ένας πίνακας μιλάει περισσότερο και καλύτερα από χίλιες λέξεις. Αυτό αποδείχθηκε από τα σκίτσα του κ. Αλή Φαρζάτ. Μέσω της δημιουργικότητάς του του, του θάρρους του και της πένας του, ε, τα σκίτσα του διεύρυναν την ελευθερία έκφραση στην ε, Συρία και σε όλο τον κόσμο. Οι πολιτικές του γελιογραφίες αντικατοπτρίζουν τα ιδανικά του. Αλή Φαρζάτ ε, ε επίθεση, βία επίθεση από τις κρατικές αρχές τον Αύγουστο. Του έσπασαν και τα δύο του χέρια. Αλλά μας έστειλε ένα μήνυμα βίντεο, δεδομένου ότι δεν μπορεί να είναι παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Σας καλώ να τον ακούσουμε. Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα πραγματικά να είμαι παρόν μεταξύ σας σήμερα κατά την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης. Δυστυχώς, ορισμένες προσωπικές ε, περιστάσεις ε, δεν μου επιτρέπουν να είμαι παρόν ανάμεσά σας. Η σκέψη μου όμως και η ψυχή μου βρίσκεται κοντά σας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου απονέμεται αυτό το βραβείο και η παρουσία μου κοντά σας, έστω και συμβολικά, εξ ε, είναι σημαντική. Όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε τα λεπτά, όσο περνάνε τα δευτερόλεπτα, έχουμε νέα θύματα στη Συρία, πράγμα το οποίο με γεμίζει πικρία. Η σκέψη μου λοιπόν ε, και τα συναισθήματά μου απευθύνονται σε αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, σε αυτούς που βρίσκονται κοντά μας, έστω και από μακριά. Όλοι αυτοί μας κάνουν μια έκκληση και μας λένε ότι η ελευθερία είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Είναι θεόσταλτο δώρο. Πριν από λίγο καιρό ρώτησα ένα φίλο μου ε, του λέω κάθε μέρα βγαίνει στο δρόμο για διαμαρτυρία, για διαδηλώσει. Δεν φοβάσαι ότι θα σε σκοτώσουν, δεν φοβάσαι το θάνατο. Ναι, μου λέει, συνεχώ το σκέφτομαι. Συνεχώ σκέφτομαι του κινδύνου που διατρέχω κάθε φορά που διαμαρτύρομαι. Αλλά αγαπητέ μου Αλή μου είπε, ξέρει πόσο σημαντική είναι η ελευθερία. Και τότε ήταν. Ε, ε, η πρώτη φορά της ζωής μου που ακούω τι σημαίνει ελευθερία. Ό,τι και να γίνει, τουλάχιστον θα έχω μιλήσει υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ελευθερίας και υπέρ της ζωής. Τουλάχιστον θα έχει ακουστεί η φωνή μου. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που μου απονέμετε αυτό το βραβείο Ζαχάροφ, που είναι μεγάλη τιμή για μένα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Τζέφρεϊ Χάρι, υπεύθυνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλους εσάς. Σας εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου. Και τώρα θα απονείμουμε τα πιστοποιητικά του βραβείου Ζαχάροφ.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 The solemn sitting is now closed. Ε, επίσημη ε, συνεδρίαση. Ολοκληρώνεται εδώ η επίσημη συνεδρίαση και θα αρχίσει αμέσως η ψηφοφορία. Voting will start immediately. Θα αρχίσουν αμέσως οι ψηφοφορίε.